εργαζόμαστε θαυμάσια. Πρόεδρος, περνάμε τώρα λοιπόν στις επεξηγήσεις ψήφων, καταρχήν όσον αφορά τις τροπολογίες για την κατάσταση στην Ουκρανία. Και ξεκινάει ο συνάδελφος κύριος Τάνοκ που μιλάει εξ ονόματος της πολιτικής ομάδας και γι' αυτό το λόγο έχει δύο λεπτά στη διάθεσή του. Η ομάδα μας θεωρεί ότι η αποτελεσματική νίκη του Πρόεδρου Ποροσέγκο, ο οποίος ε, ε, επέτυχε ε, να απελευθερώσει το Σλαβιάνσκ και ε, μπόρεσε να καταλήξει σε κατάπαυση του πυρός. Αλλά το, η, προϋπόθεση, η προϋπόθεση ήταν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να απελευθερωθούν όλοι οι όμοιροι. Αν δεν σταματήσει όμως η Ρωσία να αποσταθεροποιεί ολόκληρη τη χώρα μέσω των στρατιωτικών ενεργειών της στην ανατολική περιοχή της χώρας, τότε δεν θα πρέπει να ε, διστάσουμε να εντείνουμε τις ε, κυρώσεις. Θέλουμε ειρηνική και πολιτική λύση που να σταματήσει την ε, βία, τις απαγωγές, τον εκφοβισμό που συνεχίζουν να χαρακτηρίζουν αυτή την τραγική πρόκληση, ε, σύγκρουση. Συγγνώμη. Η λύση πρέπει να σέβεται την εδαφική ακαιρεότητα και κυριαρχία της Ουκρανίας συμπεριλαμβανομένης της Κρυμαίας, την οποία απαραδέκτως μέσω ψεμάτων ε, προσέρτηση η Ρωσία. Η πρόταση για την κυρία Μογκερίνη ω υπατή εκπρόσωπο ανησυχεί την Πολωνία και τι Βαλτικέ χώρε γιατί θεωρείται ότι η κυβέρνησή τη είναι υπέρ τη Ρωσία. Ε, μέσω τη Ιταλική Προεδρία θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τι δυνατότητε για να υπάρξει περιφερειακή σταθερότητα μετά τις, την πρόσφατη κατάληξη στην συμφωνία για σύνδεση με την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Γεωργία. Να σεβαστούμε λοιπόν τις ε, ευρωπαϊκές προοπτικές των χωρών αυτών. Ο Πρωθυπουργός Ρέντσι δεν θα πρέπει να επιχειρεί να καθησυχάσει τη Ρωσία για οικονομικούς και εμπορικούς λόγους. Γιατί ο πρόεδρος Πούτιν προσπαθεί να δημιουργήσει μια νέα Ευρωασιατική Ένωση που είναι διάδοχος της Σοβιετικής Ένωσης και προσπαθεί να προκαλέσει ε, αλυτρωτικές επιδιώξεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε Τάνοκ. Ο συνάδελφος Σογκόρ. Ευχαριστώ πολύ. Για το θέμα της ε, Ουκρανίας το βασικό είναι να αποκατασταθεί η συνταγματική ε, τάξη και η ειρήνη στη χώρα. Η αλλαγή του συντάγματος που δεν λάμβανε υπόψη τις περιφερειακές ε, διαφορές στη χώρα και δεν σεβόταν τα δικαιώματα των μειωτήτων, ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρήση της γλώσσας, ε, δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει. Εν μια δημοκρατική και κυρίαρχη Ουκρανία, όπου να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, μπορεί να επιτύχει μόνο εάν όλοι οι πολίτες έχουν τα ίδια δικαιώματα, ανεξάρτητα από το εάν αυτοί οι πολίτες χρησιμοποιούν την Ουκρανική, τη Ρωσική ή την Ουγγρική οποιαδήποτε γλώσσα. Γι' αυτό το σημαντικό είναι, τώρα που θα τροποποιηθεί το Σύνταγμα, να υπάρξει αποκέντρωση. Είναι σημαντικό επίσης οι μειονότητες και οι διάφορες περιφέρειες να παίζουν ένα ρόλο περαιτέρω στην πολιτική ζωή της χώρας. Εύχομαι κάθε επιτυχία στη χώρα αυτή. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε Σόγκορ. Παρακαλώ ορισμένους συνάδελφους να σταματήσουν γιατί αλλιώ θα τους κατονομάσω μετά την επόμενη ομιλία. Σάφορ. Σάφαζε. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, γιατί ψηφίσαμε κατά της, του κυρίου ψηφίσματος το οποίο πήρε την πλειοψηφία διότι ξεχνά το πραξικόπημα την τοποθέτηση μιας ε, επαναστατικής ε, κυβέρνησης ή την ε, ψήφο υπέρ ενός προέδρου που προεδρεύει μιας χώρας που ταλανίζεται από τον εμφύλιο πόλεμο, ώστε να συνεχιστεί ο υπεριαλισμός των ΗΠΑ. Δεν πρόκειται για ένα ψήφισμα ειρηνευτικό, αλλά για προπαγάνδα. Ευχαριστούμε συνάδελφε Σαφχάουσερ. Βίξτρομ τώρα παρακαλώ. Κυρία Βίξτρομ, μπορείτε να ζητήσετε από τη συνάδελφο να αποχωρήσει από την αίθουσα. Μπορείτε παρακαλώ να κάνετε τη συζήτηση ε, έξω. Παρακαλώ και τους επόμενους συναδέλφους που μιλάνε και θα τους κατανομάσω μετά την επόμενη ομιλία. Κέρβιν Μίκε. Ευχαριστώ. Καταψηφίσαμε διότι είναι μονομερής η αντιμετώπιση. Περίτα με αυτό το ψήφισμα ε, θέτουμε αυτούς ως αντιπάλους του Προέδρου Πούτιν. Υπάρχουν άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι ο Πρόεδρος Πούτιν θα έπρεπε να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία. Ε, απορρίπτουμε ε, μονόπλευρες επιθέσεις. Ε, Μια ισχυρή ανεξάρτητη Ουκρανία είναι προς συμφέρον της Πολωνίας. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι πρέπει να προσβάλλουμε και να δυσφημούμε ανθρώπους που δεν μας αρέσουν. Οι Αμερικανοί ψάχνουν εδώ πρόσχημα για να ξεκινήσουν ένα πόλεμο διότι βρίσκονται στα πρόθυρα της πτώχευσης και γι' αυτό το λόγο χρειάζονται ένα πόλεμο γιατί έτσι δεν χρειάζεται να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Ευχαριστώ. Να έχετε υπόψη σας ότι για τις επεξηγήσεις ψήφου δεν προβλέπονται χειροκροτήματα. Συνάδελφε Πρέντα, παρακαλώ μπορείτε να πάτε έξω να συνεχίσετε τις συζητήσεις. Η συνάδελφος Αλμπιόλ Γκουθμάν. Ευχαριστώ. Καταψηφίσαμε το ψήφισμα γιατί εμείς καταγγέλουμε τη συνεργασία των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνενοχή με την κυβέρνηση της Ουκρανίας. Η κυβέρνηση αυτή είναι αποτέλεσμα πραξικοπήματος όπου συμμετέχουν νεοναζί. Για άλλη μια φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση μπήκε στην πλευρά των οικονομικών συμφερόντων ορισμένων πολυεθνικών και των γεωστρατηγικών συμφερόντων της, ε, των Ηνωμένων Πολιτειών αντί να είναι με την πλευρά των λαών που αποτελούν την Ουκρανία. Θέλουμε μια επιτροπή έρευνας ανεξάρτητη για να διευκρινίσει το σφαγιασμό που έγινε στις 2 Μαΐου όπου στην έδρα των συνδικάτων στην Κρυμαία σκοτώθηκαν πάνω από 40 άτομα από ακροδεξιές οργανώσεις. Σε όλη την Ευρώπη πρέπει να καταπολεμήσουμε την ακροδεξιά και φυσικά και στην Ουκρανία. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος Τσίμα. Συνάδελφε Τσίμα. Συνάδελφε Τσίμα. Συνάδελφε Τσίμα. Συνάδελφε Τσίμα. Θα ήταν πολύ συμπαθητικό να παρακαλέσετε την συνάντηση που γίνεται εκεί πέρα να πάει έξω. Ο Σνάλφος Κάβα. Αν εγκρίνουμε αυτό το ψήφισμα που ξεκάθαρα οδηγεί σε χειραγώγηση, θα έχουμε επιρροές και σε πολιτισμένα έθνη που ε, ουσιαστικά καταδικάσουν τα κλίματα κατά της ανθρωπότητας και υπερασπίζονται την ειρήνη. Με την διατύπωση βλέπουμε, είπα, τους αξιωματικούς του στρατού ε, που ενδέχεται να δικαστούν θα έπρεπε ε, όμω να μην επιτρέψουμε να γίνουν αποδιοπομπή οι τράγοι, ούτως ώστε να την γλιτώσουν οι πολιτικοί. Ευχαριστούμε, συνάδελφε Κάρβερ. Στένοκα. I voted against this resolution. Εγώ καταψήφισα αυτό το ψήφισμα. Με σοκάρι που αρκετοί συνάδελφοι που προηγουμένως ε, ε, ψήφισαν αυτό το, ε, την σχέση την εταιρική με την Ουκρανία και άλλες χώρες της περιοχής για την εταιρική σχέση. Είναι πραγματικά φοβερά τα αιματηρά γεγονότα που έλαβαν χώρα τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Γιατί αφαιρέσατε το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη παράγραφο από το σχέδιο. Φτιάχνουμε τα ίδια κείμενα που βασίζονται σε άνηση μεταχείριση εκείνων στην Ουκρανία που είναι κατά της ευρωπαϊκής πορείας με αυτούς που είναι κατά. Ε, όλοι έχουν το δικαίωμα να είναι Ουκρανοί στη χώρα αυτή ε, και στο παράγραφο 8 του ψηφίσματος αυτό δεν ε, αναφέρεται. Ξεκίνησε πόλεμος, 49% των Ουκρανών έχουν αναγνωριστεί ως υποστηριχτές του καθεστώτος, ενώ 45% ότι είναι κατά. Η Ρωσία δεν αναφέρεται 33 φορές σε αυτό το ψήφισμα, ενώ η ΕΠΑ καμία. Σας ευχαριστώ κυρία Σδάνοκα, δικόπτη ο Πρόεδρος. Σας παρακαλώ ότι πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είναι δυνατόν να διαβάζετε κείμενα, διότι αν διαβάζετε ταχύτητα τα γραπτά κείμενα δεν μπορούν να παρακολουθήσουν διερμηνείς. οι επόμενοι ομιλητέ, ε, ε, εάν μιλάνε τόσο γρήγορα, θα διακοπούν από μένα γιατί δεν έχει καμία έννοια να καταλαβαίνουν μόνο οι ίδιοι αυτό που λένε. Λοιπόν, ε, τελείωσαν οι επεξηγήσει ψήφου για την κατάσταση στην Ουκρανία και θα ξεκινήσουμε τώρα τι επεξηγήσει ψήφου για την ανεργία των νέων. Πρώτο συνάδελφο Λούκε. Ο συνάδελφος Λούκε. Ανεργία των νέων να εξηγήσω γιατί ψήφισα έτσι. Καταψήφισα συγκεκριμένα γιατί το βασικό θέμα της τρέβλωσης του ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναφέρεται και που οφείλεται στο ότι το κοινό νόμισμα μειώνει την ανταγωνιστικότητα κατά τρομερό τρόπο ιδίως των κρατών της Νότιας Ευρώπης και αυτή η στρέβλωση της ανταγωνιστικότητας δημιουργεί ανεργία και κυρίως ανεργία των νέων. Είναι επίγον να αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο σκόπελο για την ανάπτυξη της απασχόλησης. Ευχαριστώ συνάδελφε Λούκε. Σόγκορ. Ευχαριστώ πολύ. Μεταξύ των νέων ε, έχουμε τρομερή ανεργία, ιδίως σε ορισμένα κράτη-μέλη. Το πρόβλημα δεν μπορούμε ούτε καν να το μετρήσουμε. Και στο μέλλον, τα επόμενα χρόνια, αυτό θα έχει και δημογραφική επίπτωση. Τα προβλήματα απασχόλησης ε, θα συνεχίσουν να επιδεινώνονται. Και είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να χρηματοδοτηθούν πλέον τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας. Πρέπει να υποστηρίξουμε οποιαδήποτε πρωτοβουλία θα βοηθήσει να βελτιωθεί η απασχόληση των νέων, αλλά χωρίς τη συμβολή των κρατών μελών αυτό δεν είναι δυνατόν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, αντιμετωπίζουν ωστόσο τρομερή γραφειοκρατία για να δημιουργήσουν θέσεις εργασία. Άρα η μείωση φυσικά θα τις διευκόλυνε. Γιατί έτσι θα μπορούσαν να τηρήσουν περισσότερο, πιο εύκολα τους κανόνες και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Ευχαριστώ. Συνάδελφο Σάντερ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, υπερψήφισα ε, το ψήφισμα διότι με 23% ανέργους ε, κάτω των 25 ετών είναι τα βασικά θύματα της ε, κρίσης και της ασθενούς ανάπτυξης αυτό οδηγεί σε δυσαρέσκεια εναντίον της Ευρώπης. Πώς να πιστέψει κανείς το ευρωπαϊκό σχέδιο όταν δεν προσφέρει καμία μελλοντική προοπτική. Η πρωτοβουλία για την ανεργία των νέων είναι μία αρχή. Όμως ε, στη δική μου εκλογική περιφέρεια αφορά μόνο σε μία περιοχή από τις πέντε. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι είναι ανησυχητική η κατάσταση με τη μακροχρόνια, όπως βλέπουμε από τις τάσεις ανεργία. Πρόκειται για διασυνοριακές περιοχές και μπορώ να σας πω ότι σε διασυνοριακό επίπεδο το δυναμικό για την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης παραμένει ανεκμετάλλευτο. Θα πρέπει να, ε, το, να το πρόγραμμα EURES, ε, να προωθήσουμε την πολυγλωσία και να ε, προωθήσουμε τα διπλά πτυχία. Θα πρέπει να επενδύσουμε στη νέα γενιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος Μελά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ψήφος μας έπρεπε να είναι αρνητική, γιατί το θέμα της απασχόλησης των νέων είναι η απόδειξη της ε, αποτυχίας της ε, διεθνούς ουτοπίας. 23% μέσος όρος ανεργίας στην Ευρώπη, 59% στην Ελλάδα ανεργία των νέων οφείλεται στο ότι είναι κακά εκπαιδευμένοι και αυτό είναι αποτέλεσμα των ε, ασυνείδητων ε, επιχειρηματιών, των ε, ακατάλληλης εκπαίδευσης. Οι νέοι μας ωστόσο είναι ένας από τους βασικούς στόχους του οικονομικού πολέμου που εξελίσσεται στην Ευρώπη και της αναγκαστικής φτώχειας και μείωση των εισοδημάτων. Εκεί συμμετέχουν ε, όλα τα θεσμικά όργανα, τα τα ταμεία έχουν χρησιμοποιηθεί λάθος, ε, δεν είναι προσαρμοσμένα στους στόχους, ε, δεν είναι λειτουργικά, ούτε η νομισματική πολιτική, ούτε η στήρα πολιτική μεταναστευτική και ο κατάλογος είναι πολύ μακρύς. Το επαγγελματικό μέλλον και το κοινωνικό μέλλον των νέων μας θα πρέπει να εξαρτάται από την εθνική κυριαρχία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Μπεγκίν. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Συνάδελφοι, παρά τις ε, προτάσεις της ομάδας μου, πρώτο μεταξύ των οποίων το αίτημα εξαίρεσης από το όριο το 30% για τις επενδύσεις ε, υπέρ των νέων δεν λήφθηκαν απόψη, ε, λόγω της θέλησης των μεγάλων κομμάτων αυτής της, ε, αυτού του κοινοβουλίου το κίνημα των πέντε αστέρων το οποίο εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή ε, αποφάσισε ε, τελικά να το υποστηρίξει. Το μήνυμα που θα ήθελα συνάδελφοι να σας δώσω αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ απλό. Πιστεύουμε πως δεν έχει σημασία από πού προέρχονται οι ιδέες ε, από τη στιγμή που είναι καλές και είναι υπέρ των πολιτών που μας ε, έφεραν εδώ για να τους ε, αντιπροσωπεύσουμε. Θέλουμε και θα εφαρμόζουμε πάντοτε αυτή την αρχή. ελπίζω τα όσα είπαν να εμπνεύσει τις εργασίες των Επιτροπών για το μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε συνάδελφοι. Είναι Ευχαριστώ. Ε, υποστήριξα ε, το ψήφισμα για την ανεργία των νέων. ούτως ώστε να συνδράμουν και εγώ για να προκύψει μία λύση για το βασικότερο πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή η υψηλή ενεργεία των νέων. Ε, στην Κροατία, όπως και σε άλλες χώρες, βιώνουμε καθημερινά τις δυσκολίες που προέκυψαν από την οικονομική κρίση και οι νέοι επλήγησαν, ε, καθώς και οι ηλικιωμένοι, σοβαρότερα από όλες τι υπόλοιπες ε, πληθυσμιακές ομάδες στην Ευρώπη. Οι ηλικίες 15 έως 24 είναι ε, η χειρότερα πληγή σε πληθυσμιακή ομάδα και αποχωρούν από την Κροατία διότι δεν έχουν καμία προοπτική και αυτό είναι το αποτέλεσμα κακών πολιτικών στα μάτια τους. Ε, ε, υποστηρίζω λοιπόν την έκκληση για την εφαρμογή της εγγύησης των νέων από τα 6 δις δεν έχει απορροφηθεί σχεδόν τίποτα από τα κράτη-μέλη και παραμένει ακέραιο το πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε. Τσινίτσι παρακαλώ Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η μείωση της ανεργίας των νέων είναι μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια καθώς πλήττει όλες τις χώρες της Ένωσης και σε ορισμένες από αυτές ε, τα ποσοστά της ανεργίας των νέων έχουν φτάσει σε απελπιστικά και ανησυχητικά ποσοστά. Πολλοί νέοι δεν βρίσκουν δουλειά και γι' αυτό το λόγο είναι υποχρεωμένοι να μεταναστεύσουν ε, σε σχέση με αυτή τη σοβαρή κατάσταση την οποία πλήττει και τη χώρα μου την Ιταλία στην νέα Κομισιόν θα ε, έχει το έργο μάλλον η νέα Επιτροπή να φτιάξει μια πολιτική που θα δημιουργήσει θέσει απασχόληση και θα σταθεροποιήσει την ανεργία. Η εγγύηση για του νέου σίγουρα βοηθά τα κράτη να αντιμετωπίσουν τη σοβαρή κρίση απασχόληση, αλλά δεν είναι και δεν μπορεί να είναι αποκλειστική και καθοριστική. Θα χρειαστούν διαθροτικέ δράσει για να ανακάμψει η οικονομία και η ανάπτυξη, ώστε να υπάρξει αύξηση τη απασχόληση. Αυτό θα συμβεί μέσω των δημοσίων επενδύσεων χωρί ε, τι πες δεν θα είναι δύσκολο να υπάρξει ανάπτυξη. Το ψήφισμα αυτό σε αυτή την κατεύθυνση κατευθύνεται και γι' αυτό το υπερψήφισα. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος Σλάιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ υπορψήφισα το ψήφισμα αυτό, αν και θα είχα προτιμήσει να ακούσω ακόμα πιο έντονα λόγια για αυτό το θέμα, το οποίο στη χώρα μου, την Ιταλία, ε, βλέπει 60% ποσοστό ανεργία των νέων ε, σε ορισμένες περιφέρειες. Η εγγύηση των νέων, ε, για τους νέους είναι δίκαιο να φτάσει μέχρι τους νέους των 30 ετών. Ακούω να λέγεται ότι θέλω να κάνω ένα παιδί, αλλά δεν βρίσκω το κουράγιο γιατί δεν ξέρω πώς θα το συντηρήσω. Επίσης θα πρέπει να ζητήσουμε να επενδυθούν περισσότεροι πόροι σε αυτό το πρόγραμμα και από αυτού νομίζω πως θα πρέπει να επιμείνουμε ε, στην Κομισιόν. Θα ήθελα να ακούσω και πιο έντονα λόγια κατά της επισφάλειας, διότι δεν είναι μόνο θέμα του πόσε θέσει απασχόληση θέλουμε να δημιουργήσουμε, αλλά να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και θέσει ποιοτικέ προ την κατεύθυνση επιτέλου ενό βιώσιμου μέλλοντο. Μια κατεύθυνση λοιπόν που είναι αυτή που πρέπει να αισθανθούμε ως ευθύνη απέναντι στις νέες γενναίες δεν ξέρω, όχι λοιπόν μόνο τι είδος θέσεων απασχόληση ε, δημιουργούμε, ένα βιώσιμο μέλλον πρέπει να δημιουργήσουμε με προσανατολισμό στο περιβάλλον, τον πολιτισμό και την έρευνα. Ο πρόεδρος διακόπτει. Ευχαριστώ συνάδελφος Λάιν. Η Κόμι. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα διότι τα στοιχεία της ανεργίας των νέων είναι πολύ ανησυχητικά και απαιτούν την απόλυτη δέσμευσή μα, την κοινή μα δέσμευση, χωρί πολιτικέ αποχρώσει. Ακριβώ επειδή πρόκειται για προτεραιότητα. Εγώ Είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι η ευκαιρία απασχόλησης για τους νέους, το να τους δώσουμε δηλαδή αυτή τη δυνατότητα, αντιστοιχεί στο να οικοδομήσουμε το μέλλον τους, αλλά και το δικό μας μέλλον. Οι νέοι είναι το πιο φρέσκο εργατικό δυναμικό της κοινωνίας μας και κυρίως αντιπροσωπεύουν το πιο γόνιμο έδαφος που πρέπει να καλλιεργηθεί μια συνεργασία, μια στρατηγική και δράσει πραγματικά ολοκληρωμένες, γιατί αυτό είναι που μας λείπει. Ολοκλήρωση ανάμεσα στα Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα είναι η καλύτερη λύση. Εντάξει, το Ταμείο Εγγύησης ε, στην Ιταλία επεκτάθηκε μέχρι τα 29 έτη, αλλά θα πρέπει να γίνουν σχετικές προσπάθειες και στα άλλα κράτη-μέλη και από εδώ θα πρέπει να ξεκινήσει η εναρμόνιση της διαδικασίας της Μπολόνια, γιατί διαφορετικά οι προσπάθειές μας θα είναι άκαρπες. Ευχαριστώ ο συνάδελφος Στεχόφσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ψήφισα υπέρ. Θα ήθελα όμως να τονίσω πως έχω σοβαρές επιφυλάξεις σε σχέση με αυτά που ακούσαμε στη συζήτηση καθώς και τη διατύπωση του ψηφίσματος. Δεν θα ήθελα βραχυπρόθεσμα να δημιουργηθούν ε, νέα προβλήματα. Πέρα από την ε, βραχυπρόθεση μάλλον ε, νέων θέσεων εργασίας, χρειαζόμαστε μία λύση συστημικού χαρακτήρα. Στην ε, Αυστρία, στη Γερμανία και στην Ελβετία υπάρχει ένα διτό, όπως αποκαλείται, εκπαιδευτικό σύστημα, ε, το οποίο έχει δώσει μέχρι στιγμής πολύ καλά αποτελέσματα. Οι χώρες οι οποίες δεν έχουν αποδώσει τη δέουσα σημασία στην μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων έχουν σήμερα ε, πολύ σοβαρά προβλήματα. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος Ζαμπόρσκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, τα μέτρα απευθύνονται σε μία μόνο ε, πληθυσμιακή ομάδα, κυρίως όταν μιλάμε για την ανεργία. Καταλαβαίνω ότι θέλουμε να θέσουμε ως προτεραιότητα την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, όμως θα έπρεπε να προκρίνουμε μέτρα που ενισχύουν την αλληλεγγύη, τη διαγενειακή. Παραδείγματο χάρη υποστήριξη των οικογενειακών επιχειρήσεων, ε, διότι όταν εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση είναι όχι μόνο αποκτούν τις απαιτούμενε δεξιότητες, αλλά μαθαίνουν ε, και την αίσθηση της ευθύνης ε, και το επιχειρηματικό ήθος από τους γονείς τους, διότι αυτό μας οδηγεί ε, στις ε, χρηματοοικονομικές κρίσεις εν τέλει. Ζητάω από την Επιτροπή να καταθέσει μια μελέτη για την κατάσταση που επικρατεί ως προς τις οικογενειακές επιχειρήσεις ε, καθώς και να εισηγηθεί η νομοθεσία για την υποστήριξη αυτών λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Σας ευχαριστούμε συνάδελφοι Ζαμπόσκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η τροπολογία υποστηρίχθηκε από την ομάδα ECR και τους συντηρητικούς. Δέχτηκε την αρχή ότι θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων, αλλά μόνο υπό όρους. Αυτό δείχνει πόσο ε, διστακτικές είναι οι απόψεις των ε, Βρετανών συντηρητικών. Είναι δηλαδή ελαφρώ ε, ευρωσκεπτική θέση. Η μασική ανεργία έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και στη Βρετανία και στην Ευρώπη. Μόνο τα εθνικά κράτη πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ε, ελέγχουν τα σύνορά του. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ούτε καν υπό όρου ελεύθερη διακίνηση αλλά μετανάστευση υπό έλεγχο με βάση συστήματα που, τα οποία θα έχουν αποφασίσει τα κράτη-μέλη και όχι ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έτσι έληξαν οι επεξηγήσει ψήφου για τα ψηφίσματα που αφορούν την ανεργία των νέων. Περνάμε τώρα στι επεξηγήσει ψήφου για τα ψηφίσματα για την κατάσταση στο Ιράκ. Ο συνάδελφο Φόικτ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, όσοι είστε εδώ ακόμη, ως ε, νεοεκλεγής με ξενίζει το γεγονός ότι ενώ η συνεδρίαση προβλέπεται μέχρι τις 2 η ώρα, ούτε 10 δεν είμαστε εδώ μέσα. Υπερψήφισα το ψήφισμα για το Ιράκ, αλλά δεν νομίζω ότι θα σημειωθεί μεγάλη πρόοδος μέσω ψηφισμάτων. Όλη η περιοχή είναι αποσταθεροποιημένη και διαρωτώ τι επέτυχε ο πόλεμος των Αμερικανών και των συμμάχων τους όταν σήμερα και πάλι υπάρχουν διώξεις όταν ε, ολόκληρες ομάδες πληθυσμού ε, ε, κακομεταχειρίζονται όταν όλη η περιοχή είναι αποσταθεροποιημένη. Λόγω της κατάστασης αυτής πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Βεβαίως ξέρουμε πόσο μεγάλα είναι τα κοιτάσματα πετρελαίου. Και δεν ξέρουμε πώ στην περιοχή αυτή λοιπόν θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι αρχές ε, της χριστιανική δύση ή της Σαρία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φόικτ. Να σας πω για να επεξηγήσω την κατάσταση. Οι επεξηγήσει ψήφου γίνονται μετά την ψηφοφορία. Οπότε μένουν μόνο εκείνοι που θέλουν να επεξηγήσουν την ψήφο του. Αυτό το τμήμα τη Ολομέλειας δεν έχει ως στόχο να ακούσουν όλοι οι συναδέλφοι. Πρέπει να το καταλάβετε όλοι αυτό. Γι' αυτό το εξηγώ. Λόγω των αντιδράσεων που υπήρχαν. Πρέπει να σας εξηγήσω ότι ούτε στο Εθνικό Κοινοβούλιο, ούτε στα κοινοβούλια, ε, το Κοινοβούλιο της Ένωσης δεν συνηθίζεται να υπάρχουν αντιδράσεις από το θεωρείο. Από τα θεωρία των ε, θεατών των επισκεπτών. Ο κύριος Χάπερ δεν είναι εδώ, οπότε έληξε να ψήφου για το Ιράκ. Περνάμε σε επεξηγήση ψήφου για την ε, κλιμάκωση βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Ένα άνθρωπος θέλει να πάρει το λόγο, ο Σάλφος Φόικτ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Υπερψήφισμα το ψήφισμα αυτό, αλλά δεν πάει αρκετά μακριά. Χθες στη συζήτηση ιδιαίτερο ο κύριος Λάμστορφ, αναφέρθηκε το δικαίωμα άμυνας του Ισραήλ. Πρέπει να το συμπληρώσουμε αυτό λέγοντας ότι μια χώρα όπως η Παλαιστίνη που είναι υποκατοχή εδώ και δεκαετίες που έχει χωριστεί σε τμήματα, που έχει διχοτομηθεί όπου έχει ε, οικοδομηθεί ένα τείχος για να την περιορίσει όπου υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες σε άλλες διπλανές χώρες έχει και αυτή η χώρα δικαίωμα να αμήνεται Επιθυμώ όμως να επανέλθει σύντομα στην περιοχή η ειρήνη και εμείς με τα ψηφίσματά μας και ίσως με πιο ενεργή πολιτική να μπορέσουμε να συμβάλλουμε. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη πάντα τα συμφέροντα και των δύο πλευρών και όχι μόνο της μίας. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Οπότε έληξαν επεξηγήσεις ψήφου και λίγοι και η ε, εβδομάδα Ολομέλειας. Εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους που είναι ακόμη εδώ καλή επιστροφή, καλές διακοπές με ανάπαυση. Ευχαριστώ επίσης τις υπηρεσίες μας εδώ, δεξιά-αριστερά, πίσω μου. Ιδιαίτερα ευχαριστώ και τους διερμηνείς της καμπίνες. Νομίζω ότι και εσεί έχετε κερδίσει με την εργασία σας ε, διακοπέ. διακοπές. Ο Σάρφο Μπάλι είχε δει το λόγο για διαδικαστικό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήταν πάρα πολύ ευγενικό που μου δίνετε το λόγο. Για μένα είναι ε, λυπηρό να μιλάω σε τόσο άδεια αίθουσα όπως είπε και ο συνάδελφος. Εγώ θα ήθελα να θυμίσω ότι εμείς είμαστε εδώ, πληρωνόμαστε έδρα από τους ε, φορολογόμενους για να κάνουμε μια δουλειά. Και αν πρέπει να την κάνουμε αυτή τη δουλειά θα πρέπει να την κάνουμε με συνέπεια και ικανότητα. Και έχω την εντύπωση ωστόσο ότι δεν υπάρχει σεβασμός για αυτή την εργασία από πλευρά των συναδέλφων. Γιατί είδα πραγματικά δηλώσεις που γίνονται σε πλήρες ε, χάος και εσείς είπατε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πάνε να πάρουν το αεροπλάνο. Μα δεν μας πληρώνουν για να πηγαίνουμε να παίρνουμε τα αεροπλάνα, αλλά για να εργαζόμαστε με μεγάλη σοβαρότητα. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Είστε νέος ε, συνάδελφε. Ε, δεν σας πήρα το λόγο παρά το ότι δεν πήρατε το λόγο για διαδικαστικό. Ήταν μια γενική πολιτική δήλωση. Ε, πληρωνόμαστε για να τηρούμε τους κανόνες, ξέρετε. Θέλει κανεί ε, άλλο το λόγο για διαδικαστικό. Μόνο για διαδικαστικό παρακαλώ. Μόνο διαδικαστικό παρακαλώ. Προεδρεύσατε με εξαιρετικό τρόπο. Προέδρε, συγχαρητήρια. Νομίζω ότι ο τελευταίος ομιλητής δεν ήταν πολύ δίκαιος, γιατί υπάρχουν και βουλευτές που δεν έχουν άλλη επιλογή, μόνο τώρα έχουν αεροπλάνο για